Señor presidente. Se reanuda la sesión. Tienen... Να ξεκινήσουμε εκ τη συνεδρίαση. Έχετε ουσιαστικά τα πρακτικά στη διάθεσή σας της χθεσινή συνεδρίαση. Αν κάποιος ε, θέλει σχετικά το λόγο, παρακαλώ. Αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που έχει να κάνει με μια δήλωση της